Λοιπόν, ε, να τα ξαναπώ ότι από την αρχή τη ε, καρδιά μου στο Κοινοβούλιο ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Βλέπω θετικά στοιχεία στο σύστημα ε, εμπορίας, εμπορία ανταλλαγή πιστώσεων ρήπων του άνθρακα, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί για κάποια άλλα πράγματα. Η ευρωπαϊκή πολιτική κλίματος έχει ένα πολύ ψηλό τίμημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία πανάκριβη, την πλέον ακριβή μονομερή πολιτική κλίματος στον κόσμο που α, οδηγεί σε μείωση της εργασίας και τιμωρεί ακόμα και καθές μορφές εργασίας. Και όταν μιλάμε για το ETS θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε να το λέμε. Οι τελευταίες, οι πλέον προσφορέ έρευνες λένε ότι η, η φυστάμενη πολιτική ούτε καν μειώνει τις εκπομπές. Τι εννοώ. Αν λάβουμε υπόψη την κατανάλωση και τις συνολικές εκπομπές της Ένωσης, τότε έχουμε αύξηση των εκπομπών. Ενώ οι εκπομπές που οφείλονται στην παραγωγή, ναι, πράγματι μειώθηκαν λόγω του ETS. Περίεργο λοιπόν είναι ότι οι εκπομπές που βασίζονται στον κατασκευαστικό κλάδο δραματικά αυξήθηκαν. Αυτό δείχνει ότι αποτύχαμε, αποτύχαμε δραματικά. Γιατί ουσιαστικά μεταφέραμε τις εκπομπές των ρήπων σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου παράγουν λιγότερο καθαρά. Και ταυτόχρονα παρήγαμε μεγάλη ανεργία στην Ευρώπη. Ε, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και αυτό αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Όταν μιλούμε για ε, προστασία ε, του κλίματος, ε, να μην νομίζουμε ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο θα πρέπει να ασχολούμαστε όχι μόνο με την παραγωγή εκπομπών, αλλά και με την κατανάλωση. Γιατί αυτές είναι οι δύο μορφές εκπομπών ρήπων. Γι' αυτό δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί εστιάζουμε σε αυτό το μηχανισμό ETS εις βάρος ουσιαστικά του απότερου στόχου μια πολιτική παρέμβαση στις τιμές μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα οικονομικά αποτελέσματα και να υπονομεύσει ε, καταλυτικά την οικονομική ανάκαμψη. Ήδη προβλέπεται ότι μεγαλύτερη Χρήστε ενέργεια στην Ευρώπη μπορούν να δουν την χρήση ενέργεια να αυξηθεί κατά 1,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, 3% αύξηση ετησίω ε, προβλέπεται με αυτό τον ε, ρυθμό. Γι' αυτό ζητώ μια διευκρινιστική τροπολογία. Είναι μήνυ τροπολογία, όπως λέει η Κομισιόν. Ώστε η Κομισιόν να μπορεί να ελέγχει την αγορά, αλλά όχι να τη χειραγωγεί την αγορά, γιατί αυτό η χειραγώγηση της αγοράς θα οδηγήσει σε μεγάλη ανασφάλεια. αλλά ακόμα και αν γινόταν μόνο μία φορά αυτό και πάλι το τελικό κόστος για τους ιδιώτες, τα νοικοκυριά δηλαδή, αλλά και τις βιομηχανίες θα ήταν πολύ υψηλότερο. Και όλα αυτά σε μια στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία πασχίζει να βγει από την κρίση και να βρει μια σταθερότητα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε θετικά κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα τεχνολογικά ευρήματα για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να μην κάνουμε το αντίθετο. Η... Απευθύνω λοιπόν μια έκκληση στους ελιστές φίλους να το ξανασκεφτούν. Θέλετε ανάπτυξη. Ε, αφήστε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Μην ε, του χτυπάτε στα πλέον ευάλωτα του σημεία. Άκουσα να λέτε ότι θα δοθεί μια προτεραιότητα στον άνθρακα αφήνοντας το σύστημα ETS ως έχει. Οι εταιρείε ενέργεια δεν χρησιμοποιούν τον άνθρακα λόγω τη χαμηλή τιμή, αλλά λόγω χαμηλή τιμή του κάρβουνου. γιατί έχουμε πολύ φθηνέ εξαγωγέ άνθρακα στην Ευρώπη. Το backloading τελικά δεν επηρεάζει τις τιμές, είτε το αποδεχτούμε είτε το απορρίψουμε. Και έχουμε δύο αλλαγές ε, να λάβουμε υπόψη, ότι το ETS το σχεδιάσαμε για άλλη εποχή. Ούτε ενεργειακό πρόβλημα είχαμε, ούτε οικονομικό πρόβλημα, οικονομική κρίση είχαμε. Ήταν σχεδιασμένο σε μια εποχή ευημερία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τη σημερινή κατάσταση και να δούμε και την κατάσταση ενεργειακού εφοδιασμού και στις ΙΠΑ την επόμενη πεντακονταετία, καθώς εκεί αναμένεται ότι οι ενεργικέ τιμές να είναι χαμηλές στο 1 τρίτο των ευρωπαϊκών τιμών και οι τιμές ηλεκτρισμού θα είναι σταθερές επίσης, ενώ αντίθετα και το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη θα αυξάνουν συνεχώς διευρύνοντας το ανταγωνιστικό αυτό χάσμα με τον μεγάλο μας ανταγωνιστή της ΕΠΑ. Άρα θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η λύση σήμερα. Το backloading θα βοηθήσει σε αυτό το πρόβλημα. Όχι, λέω. Γιατί το backloading δεν θα οδηγήσει σε πραγματικές λύσεις αλλά μόνο σε αύξηση του κόστους της ενέργειας σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Αυτό λοιπόν το μέτρο του backloading μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ανθρακά από 5 στα 10 και σε 15 ευρώ, αλλά όχι ποτέ σε 50 ευρώ που είναι το κατόφλι για πραγματική αλλαγή ε, σε πηγή ενέργειας, το power switch. για να αλλάξουν την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν οι εταιρείε και να χρησιμοποιήσουν τον άνθρακα και όχι το κάρβουνο, συγγνώμη, το κάρβουνο και όχι ε, το αέριο, θα πρέπει οι τιμές να είναι πολύ διαφορετικές και να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο χάσμα. Οι τιμές σήμερα, όπως προβλέπονται, είναι μη βιώσιμες. Ειδικά μέσα στην εποχή της κρίσης. Το backloading λοιπόν δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε μέτρα που να μπορούν να μας επιτρέπουν να κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις στο μέλλον. Μόνο έτσι θα έχουμε μια κάποια ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το απαραίτητο κίνητρο για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Αυτό λοιπόν το μέτρο του backloading δεν πρόκειται να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση πολλοί λόγοι για τους οποίους η δικιά μας ομάδα δείχνει τέτοιους δισταγμούς έναντι των προτάσεων της Κομισιόν. Και οι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο, θα πούν περισσότερα. Φοβούμεθα ότι ούτε είναι κατάλληλη στιγμή, ούτε η κατάλληλη πρόταση. Το ETS πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργήσει χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Το ETS θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο τεχνολογικά ουδέτερο με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να είναι αποτελεσματικό οικονομικά και πρακτικά. Λυπούμε αν το πω, αλλά θα το πω, ότι ε, η κερδοσκοπία ήδη, ε, όπως και οι εικασίες, έχουν επηρεάσει πολύ αρνητικά το όλο σκηνικό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κρίς Ντέιβις. Και εγώ εργάζομαι από την αρχή όταν δημιουργήθηκε αυτό το σύστημα με το ETS. Η κυρία Κοχόλ έχει απόλυτα δίκιο με την έννοια ότι πάντοτε ήταν ακόλουθη ε, στα λεγόμενα της. Από τα πρώτα χρόνια πάντοτε την ίδια γραμμή κρατούσε. κάποιες φορές ε, δεν μπορεί να θυμηθεί, ε, δεν κανείς ότι ήταν από το έλκο εισηγητής που προωθούσε το ETS. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε πρώτα και μέτρα για να ενισχύσουμε ε, το σύστημα ETS και θυμάστε και τη σχετική ψηφοφορία πέρυσι με 400 ψήφους υπέρ, ζητώντας την Κομισιόν να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο πιστώσεων δεν κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Μιλάμε για το backloading. Είναι πραγματικά ένα ασήμαντο ποσοστό στο όλο σύστημα και έχει γίνει τέτοιες έντονες συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Εκπληκτικό. Γιατί φαίνεται ότι χρησιμοποιείται σαν δούριο ύπο για να επιτεθεί όχι για να γίνει επίθεση όχι μόνο στο ETS, αλλά οτιδήποτε κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος. Και δεν άκουσα τίποτα από τη συνάδελφο για εναλλακτικέ. Δηλαδή πώς βλέπετε το μέλλον. χαμηλέ τιμέ ενέργεια θέλετε. Ωραία. Πώς θα γίνει αυτό με το κάρβουνο, δηλαδή θα ε, κινούμεθα στο μέλλον. Αν ο άνθρακα θα στα 4 ε, ευρώ, δεν ξέρω πώ θα μπορέσετε να υποστηρίξετε τέτοιου είδου υποδομέ. Ποιο είναι το όραμά σα, μακροχρόνια το όραμά σα. Αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε. Όταν ε, είχαμε τα πρώτα βήματα του ETS, οι τιμέ ήταν 30 ευρώ τον τόνο. Περιμέναμε πριν την ύφεση να αυξηθούν αυτέ οι τιμέ. Τώρα είμαστε στα χαμηλότερα α, ιστορικά. Περίπου 4 ευρώ τον τόνο. Κάπου λέει το κείμενο ότι οι επενδύσεις ε, δεν υπάρχουν γιατί περίμενα 40 και 50 ευρώ. Μα μου έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει ο κόσμος. Α, όταν η Κομισιόν έκανε την πρόταση για το backloading, α, δεν προσπάθησε να κάνει ουσιαστικέ αλλαγέ στο ETS, αλλά να αντιμετωπίσει την κρίση ώστε να μην καταρρεύσει η αγορά εν γέννη. Ξέρουμε ότι έχουν ε, καταργηθεί, ακυρωθεί, συγγνώμη, μάλλον πολλέ δημοπρασίε. και για μας είναι σημαντικό αυτό. Ε, ε, εμείς και το Συμβούλιο έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θέλουμε να λειτουργήσει και βλέπουμε να μην λειτουργεί. Και βλέπουμε ε, απώλεια οποιασδήποτε επιθυμίας επενδύσεων. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον ζωντανό το ETS. Ποιες είναι οι συνέπειες του μέτρου αυτού Ακούσαμε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ε, διάφορα σχόλια από τον Boy ότι αν περάσει το backloading τότε μπορεί να φτάσει η τιμή 8 ευρώ τον τόνο. Εκείνη τη στιγμή ήταν 7 ευρώ τον τόνο. Εντάξει, δεν φοβήθηκε κανείς. Αν τώρα δεν περάσει το backloading τότε θα πέσει η τιμή στα 5 ευρώ τον τόνο. Αλλά και εκεί την πάτησε γιατί ε, έπεσε ακόμη περισσότερο. Φτάνει σχεδόν τα 3 ευρώ τον τόνο. Ακούσαμε από όσους είναι κατά της πρότασης για το backloading ότι η Κομισιόν ε, ξεπερνά τα εσκαμμένα και ξεπερνά τις ε, εξουσίε τη. Μα μέσω της συναπόφασης ε, η Κομισιόν δεν ξεπερνά ποτέ τα όρια της. Και άκουσα τα επιχειρήματα ότι η Κομισιόν είναι ο ρυθμιστής του ETS. Μα άρα λοιπόν δεν χρειαζόταν καν να υποβάλει αυτή την πρόταση. Γιατί έχει η ίδια την εξουσία βάσει της συνθήκης να λειτουργήσει ρυθμιστικά και να ορίσει το χρονοδιάγραμμα αυτών των δημοπρασιών. Πάντως ήρθε και επέβαλε νομοθετική πρόταση. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να παρέμβουμε στην αγορά και ότι χειραγωγούμε την αγορά με αυτόν τον τρόπο αλλά η κυρία Κόχορ παρούσα δεν ήταν όταν η κυρία Βάλστρομ ως επίτροπος ε, παρουσίασε την πρότασή της και τι μας είπε, ότι κάνοντας μαθαίνουμε και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Άλλε χώρε στον κόσμο μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ε, δημιουργούν δικά του συστήματα ETS, μαθαίνουν από την εμπειρία τους. Ε, και εμείς δεν πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία μα. χρειάζεται κάποιε φορέ να ε, τρανταχτούμε από κακές εμπειρίες πριν καν καταρρεύσει το όλο σύστημα, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Τώρα για την αβεβαιότητα και τις επενδύσεις. Τι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στους επενδυτές όταν δεν υπάρχει όραμα για το μέλλον. Τι μας λέτε εσείς και η εκλογή σας. Αν θέλουμε ένα μέλλον με χαμηλή χρήση άνθρακα, χρειάζεται δύναμη σήμερα και κίνητρα για να κινηθεί η αγορά προς επενδύσεις με χαμηλή χρήση άνθρακα. Το backloading δεν θα το κάνουν αυτό. Το backloading ουσιαστικά αλλάζει το χρονοδιάγραμμα των ε, δημοπρασιών για να μην καταρρεύσει το όλο σύστημα των, ε, της των πιστώσεων. είναι μια πολύ μικρή πρόταση που δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στην πρόταση. Παρακαλώ λοιπόν, απευθύνω αυτή την έκκληση να την εγκρίνουμε την πρόταση γιατί δεν θα επηρεάσει τίποτα ουσιαστικό. Ούτε τις επενδύσεις, ούτε την κερδοφορία των βιομηχανιών έντασης ενέργειας. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είπατε ότι οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεκαθίσατε άλλο σε άλλες χώρες. Όχι όλοι, όχι. Άλλοι μένουν εδώ. Άλλοι που φεύγουν το κάνουν γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε καμία περίπτωση τις τιμές σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά μας είπατε ότι οι τελευταίες έρευνες ε, τις οποίες δεν μας αναφέρετε ποιες είναι, ότι πρόσφατα ενεργειακές ε, επιχειρήσεις κάνουν κέρδος. Πού? Εγώ σας ρωτώ, ακόμα και οι αερομεταφορείς ακούστηκε πρόσφατα ότι κάνουν τέτοια κέρδη. Όχι, είναι μύθος όλα αυτά. Όποιος αλλάζει την έδρα του σε μια άλλη χώρα του κόσμου, δραγκαστικά άξαν το κέρδος. Και εγώ θέλω να τους κρατήσω όλους εδώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ. Chris Davis. Ο Μπάς Άικαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσα εδώ να ξεκινήσω μια ιδεολογική συζήτηση για την κλιματική κρίση και τι πρέπει να γίνει. Θα μπορούσα να ξεκινήσω μια συζήτηση για τα ε, πόσες επιχειρήσεις έβγαλαν χρήματα αυτή τη στιγμή από τις ε, ε, από τα επιδόματα θέλετε, που λάβανε στη δεύτερη, εμπορία, στη δεύτερη περίοδο εμπορία. Ε, μια χώρα που είναι πολύ φιλόδοξη ε, στην ενεργειακή μετάβαση και πιο ανταγωνιστική οικονομία στην Ευρώπη, η Γερμανία. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι να αναφερθώ στην Αυστραλία που έχει ένα σύστημα με την τιμή των 17 ευρώ. Επομένω, όσοι λένε ότι είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, εγώ θα σα έλεγα πηγαίνετε στην Αυστραλία, αν θέλετε να είστε πραγματικά φιλόδοξοι. Θα μπορούσα να τα, να τα πω όλα αυτά και να ζητήσω μέτρα. Όμω έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Έχει αλλάξει το κέντρο βάρου τη συζήτηση. Και πραγματικά διαρωτώ με αν οι συνάδελφοι έχουν επίγνωση του γεγονότο ότι έχει αλλάξει αυτή η συζήτηση. Δεν μιλάμε πλέον για αυτά τα θέματα. Μιλάμε για τη διάσωση του ESTS. Αυτό είναι εδώ το θέμα. Η τιμή έχει, περάσει, έχει πέσει κάτω από τα 5 προ τα 4 πάει, πέφτει κάθε μέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε δημοπρασία 4 εκατομμυρίων ε, ε, τέτοιων δικαιωμάτων στη Γερμανία που ακυρώθηκε γιατί δεν υπήρχε κανένα αγοραστή. Ο μοναδικό λόγο που υπάρχει ακόμα τιμή είναι επειδή υπάρχουν κάποιε επενδύσει, Κάποιοι επενδυτέ που πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί και να λειτουργήσει το σύστημα, αλλά και αυτοί μειώνονται κάθε μέρα. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν, περί του μέλλοντο του ETS. Και όσοι συνάδελφοι λένε ότι εγώ είμαι κατά του backloading, έχω το εξή απλό ερώτημα για αυτού. Είστε υπέρ του ETS, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν απλώ θέλετε να το ξεφορτωθείτε, όπω η κυρία Κόλλα, κανένα πρόβλημα. Απλώ πείτε το όμω. Μην μου λέτε αυτέ τι ανοησίε και αυτά τα επιχειρήματα για το τι κάνουμε στην αγορά και τα αν τη Εξ αρχή γίνεται αυτό, εφόσον έχουμε τιμή για τον άνθρακα. Ε, αυτή είναι η ουσία του συστήματο. Μην μου λέτε λοιπόν αυτέ τι ανοησίε. Πείτε μου ειλικρινά, εγώ είμαι κατά του ETS. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε μια ξεκάθαρη συζήτηση. Όμω μετά θα ήθελα να αναφερθώ στου συναδέλφου ε, τη κυρία Κόλλερ που ήταν υπέρ του ETS και πάλευαν υπέρ του ETS. Τώρα πράγματι ε, ακολουθείτε κατά του backloading ή θέλετε να παλέψετε για το ETS. Γιατί αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή απλώ κερδίζουμε χρόνο πριν πραγματικά καταρρεύσει εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτή την πρόταση. Από πλευρά πρασίνων το backloading δεν είναι τίποτα. Θα ανέβει τιμή στο 5, στο 6 αν είμαστε τυχεροί. Ε, να αναβάλουμε τη συζήτηση προ τον επόμενο επίτροπο, οποίο και να είναι αυτό. Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα, απλώς αναβάλουμε τη συζήτηση. Και αν μείνουμε στο backloading το πρόβλημα θα υπάρχει και το, το 2016-2017. Γιατί τότε θα πλημμυρίσει, αν θέλετε, το σύστημα. Επομένω για αυτό το πράγμα μιλάμε, για, το, ε, για να κερδίσουμε χρόνο. Εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω, όπως και η Βρετανική κυβέρνηση, με τα διαθετικά μέτρα, γιατί θέλω παραπάνω. Ναι, αυτή την ιδεολογική συζήτηση να την κάνουμε. Πώς θα σώσουμε το σύστημα. Αυτά να μας πούνε, οι συνάδελφοι. Ίσως δεν είναι υπέρ του παραμερισμού του ΣΕΤΑ αλλά πείτε μου τι θέλετε. Ή να το εγκαταλείψουμε, αν αυτό θέλετε. Ε, αναφερθήκατε στο Συμβούλιο. Εκεί η Γαλλία είναι υπέρ, η Ισπανία, η Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να πάει παραπέρα. Ο Ιρλανδό Υπουργό Θε είπε ναι, θέλουμε ε, συζήτηση για το αν επιθυμούμε να διατηρηθεί το ETS ε ή όχι. Το Συμβούλιο <laughs> ουσιαστικά έχει ξεπεράσει το Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι απίστευτο. Ε, πριν παλιότερα ήμασταν μπροστά σε αυτή την πάλη και τώρα έχουμε μείνει πίσω. Το Συμβούλιο τώρα μόνο μένει να δει τι ακριβώς θα κάνει η Γερμανία. Τότε η Γερμανία θα είναι υπέρ, τότε θα περάσει. Και τότε το Συμβούλιο θα είναι υπέρ. Και εμείς εδώ συζητούμε χαζά επιχειρήματα. Είναι πρόβλημα του Κοινοβουλίου και είναι κάτι που με λυπεί πολύ. Γιατί από πλευρά Πρασίνων θα μπορούσαμε να πάμε πολύ παραπέρα. Αλλά ούτε καν αυτή τη συζήτηση δεν κάνουμε. Τελευταία παρατήρηση. Εάν οι συνάδελφοί μου είναι ειλικρινεί και πούνε δεν θέλουμε το ESDS, εντάξει, κανένα πρόβλημα να δούμε όμως και τον κατάλογο ε, carbon leakage, ε, διαρροής άνθρακα που έχει σχεδιαστεί με την τιμή των 30 ευρώ. Πρέπει να ε, αναθεωρηθεί λοιπόν. Αν σκοτώσουμε ε, το σύστημα ETS, τότε να ξεφορτωθούμε και, αυτή, και αυτό το κατάλογο που βασίζεται στα 30 ευρώ. Γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, βοηθάμε τι επιχειρήσει από όλε τι πλευρέ, του δίνουμε χρήματα καινοτομία ε, για την χαλιβουργία, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή ε, εργάζονται επί τη καινοτομία με ευρωπαϊκά χρήματα, ε, έχουν λάβει λοιπόν κονδύλια από εκεί για να αντισταθμίσουν τον ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε τον κατάλογο με τα 30 ευρώ, τα έχουμε όλα. Ας τα διαγράψουμε και αυτά τότε ας κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ή απλώς στηρίξτε αυτή την, αυτό το απλό ζήτημα να κερδίσουμε χρόνο και μετά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Χρειαζόμαστε χρόνο όμως, αλλιώς θα καταρρεύσει το σύστημα και να θυμάστε ότι είστε και εσείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Μάρτιν Κέλλερμαν. Ευχαριστώ, Ματιάς που μου δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχω στη συζήτηση. Ε, φαίνεται ότι περισσότερο αφορά ε, τις μεθόδους, τους τρόπους, ε, παρά τα ωφέλη της συγκεκριμένης πρότασης. Πριν περάσω λοιπόν ε, στην ε, πρόταση, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στη συζήτηση. Ε, με έχουν προβληματίσει ε, ο Chris Davis και ο Μπάς Έκοτς στις ε, παρεμβάσεις τους. Αν αυτή η πρόταση είναι πραγματικά μια χάσιμο χρόνου, τότε γιατί ε, ασχολούμεθα με αυτό το θέμα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι και τόσο αδιάφορο. Θα θα είναι σημαντική η πρόταση, γι' αυτό και έχει κατατεθεί. Αν και οι ενθουσιώδεις υποστηρικτέ πρέπει να μα εξηγήσουν ε, γιατί είναι τόσο ενθουσιώδεις. Διακόπτη συνάδελφο και λέει ότι απλώ κερδίζουμε χρόνο. Λοιπόν, και πάλι για να απαντήσω και στον Βάσ και στον Κρι για την διαρροή άνθρακα. Είναι μια περισσότερο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντο συζήτηση. Αλλά είναι ένα πραγματικό γεγονό στη δική μου περιφέρεια. Ε, αναφερθήκατε στην παραγωγή αλουμινίου. Είχαμε μια πολύ μεγάλη ε, τέτοια εγκατάσταση στην βόρεια βορειοανατολική Αγγλία με 400 υπαλλήλου ε, σε μια εποχή μεγάλης ανεργίας και έκλεισε φέτος εξαιτία του ETS και εξαιτία της, ε, ε, οδηγίας περί μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης. Και πού πήγε, πού μεταφέρθηκε αυτή η εγκατάσταση, αυτό το εργοστάσιο, στην Ινδία, στην Κίνα, χαμηλής ε, παραγωγής, όχι, στον Καναδά πήγε. με υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, υψηλότερου μισθού, υψηλότερο κόστος παραγωγής από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ε, στον, ε, στην τιμή του άνθρακα και υψηλής έντασης οικονομία. Είδαμε λοιπόν ότι με μεγάλη επιτυχία μεταφέρθηκαν ε, εκατοντάδε θέσει εργασία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε πολλέ άλλου κλάδου τη βιομηχανία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε να, να σηκώσουμε το βάρο αυτή τη απόφαση, να πληρώσουμε το τίμημα. Όμω ε, και πολλέ από αυτέ τι νέε πράσινε βιομηχανίε στηρίζονται στι κρατικέ επιδοτήσει. Και αν θέλετε ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό είναι το μέλλον, εντάξει, ε, προωθήστε αυτό το επιχείρημα. Όμω ε, μην ε, χρησιμοποιείτε το επιχείρημα τη διαρροή άνθρακα, γιατί δεν είναι σχετικό. Περνώ τώρα στα υπέρ αυτή τη πρόταση. Τα έχουμε συζητήσει επί μακρόν βέβαια, τα έχουμε πει όλα, όμως ήταν ένας μηχανισμός της αγοράς έτσι είχε δημιουργηθεί ε, και στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είχε ζητηθεί πρώτη φορά τα είχαμε πει αυτά και ο Κρίς είχε δίκιο. Το τότε Επίτροπο είχε πει ότι η Επίτροπος είχε πει ότι πράγματι ε, ζούμε και μαθαίνουμε, έτσι λοιπόν από τα λάθη μας τα μάθουμε. Όμως ε, λέγαμε ότι η Ευρώπη ηγείται του κόσμου και ότι όλοι ανησυχούσαν τόσο πολύ για, τις, για την κλιματική αλλαγή που όλοι θα μας ακολουθούσαν. Όμως βλέπουμε ότι δεν το πράττουν. Ε, Κάποιε φορέ, λένε, αν θέλετε, ισχυρίζονται ότι ακολουθούν τι ίδιε αρχέ, όμω εν γέννη δεν ε, το πράττουν. Ακούσαμε και τα θερμά λόγια εντό εισαγωγικών του Προέδρου Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα και θα δούμε τι θα γίνει και αν είπα, θα αναλάβουν κάποια δράση. Γιατί από τι δικέ μου συζητήσει ε, με γερουσιαστέ ε, στι ΣΥΠΑ δεν υπάρχει παραμικρή πρόθεση να γίνει κάτι. Βεβαίω η οικονομία της, των ΗΠΑ αναπτύσσεται εξαιτία της χαμηλής τιμής ε, του συστολιθικού αερίου. Ε, Βεβαίω, η Επιτροπή ήθελε ένα μηχανισμό που θα βασίζεται στην αγορά, ήθελε να λειτουργήσει. Βεβαίω, έχει πέσει τόσο πολύ η τιμή του άνθρακα. Έχω 5,60 ήταν η τιμή που ξέρω εγώ. Βέβαια, ακούω σήμερα ότι έχει πέσει παρακάτω. Αλλά το σύστημα δεν λειτουργεί καλά, δεν ε, παράγει τα όσα θέλαμε. Όμως ε, η ύφεση οδήγησε σε αυτή την μείωση της τιμής γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση αδειών. Αποδεχόμεθα ότι δεν λειτουργεί σωστά ε, βάσει της αρχικής πρότασης που είχε υποβληθεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει και τόσο σημαντική διαφορά και θα βελτιώσει την κατάσταση η συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Διαδικαστικό από την κυρία Κορόλα. Ναι, ήθελα μόνο να διορθώσω ε, ένα λάθος μόνο. One mistake. Διαδικαστικό μου είπατε. Ε, διαδικαστικό ζητήσατε. Ποια είναι η σωστή διαδικασία, λέει η κυρία Κορόλα. Ο κύριος Σιμάνσκι. Πώς μπορώ να διορθώσω κάτι που υπόθηκε για μένα και το οποίο είναι λάθος. Στην Ολομέλεια Γενικά μπορεί κανείς να πει αν υποθεί κάτι λάθος. Ε, ναι, έχουμε την μπλε κάρτα, λέει ο πρόεδρος. Ε, ε, έχετε κάτι διαδικαστικό? Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Ποτέ δεν είπα ότι... ότι θα πρέπει να μάθουμε κάνοντας. Ο κύριος Βίκμαν το είπε από την ομάδα μας. Ωραία τέλος, λέει ο πρόεδρος. Τέλος, δεν είμαστε παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν κάνοντας, αλλά εμείς δεν είμαστε παιδιά. Προτείνω να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Εάν υπάρχει κάποιο διαδικαστικό, μπορούμε να το επιτρέψουμε, αλλά τίποτα παραπάνω, διότι έχουμε πολλούς συναδέρφους ε, στη, στον κατάλογο ε, και ε, δίνω τον λόγο στον κύριο Τσιμάνσκι. Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι στην αρχή της παρέμβασής σας μιλήσατε για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, χωρίς καν να ρωτήσουμε κατά πόσον χρειάζονται να γίνουν αλλαγές. Γιατί δεν είναι μόνο το πώς θα γίνουν αλλαγές, αλλά και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, σε σχέση με αυτή την πρόταση και πρέπει να ακουστούν όλες οι προσεγγίσεις. Εγώ συμφωνώ με όσους είπαν ότι αυτή η μείωση που θέλουμε να επιτύχουμε είναι σημαντική, είναι πραγματικά ασήμαντη εντελώ. όπως είπε και η προλαλή α, πραγματικά, αν είναι κάτι ασήμαντο το θα επιτύχουμε, γιατί πραγματικά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία το σύστημα θέλει να δημιουργήσει μηχανισμούς τέτοιους ώστε να επηρεάζονται οι παραγωγοί ως προς την παραγωγή τους ε, να αλλάξει η δομή παραγωγής ενέργειας. Αυτό δεν είναι το νόημα αυτού του ETS. Τώρα, εδώ μιλάμε για ουσιαστικά για ένα lifting, ε, για κάτι πολύ δευτερεύον, για μια μικροαλλαγή στο σύστημα και ρωτώ ποιο είναι το νόημα. Δηλαδή όποιο διαφωνεί επίσης δεν πρέπει αμέσω να στιγματίζεται με κακές προθέσεις κτλ. Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων άρχισε να επιτίθεται στην κυρία Κόχαλα και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει έτσι η συζήτηση. Όλοι, όλοι συμφωνούμε ότι η μέση δικτύου του άνθρακα συνδέεται άμεσα με το μέλλον του πλανήτη μας, πράσινο ή όχι. Η κυρία Κοχάλα είπε ότι είναι ένα πολύ σχηδές πρόβλημα, ένα περίπλοκο πρόβλημα και δεν μπορεί έτσι απλά να κάνουμε τη συζήτηση ναι ή όχι σε ένα μηχανισμό. Υπάρχει και ε, η διάσταση της επιχειρηματικότητας, η οικονομική διάσταση, τόσες διαστάσεις. Ακούσαμε και παραδείγματα από συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες ότι ε, το εργοστάσιο αλουμινίου δεν μπήκε σε τρίτη χώρα του κόσμου αλλά μπήκε στον Καναδά. Να ένα ωραίο παράδειγμα στην Πολωνία, στη χώρα μου, αλλά και στην Ισπανία και στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι τεράστιο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα εργατικά χέρια στη βιομηχανία. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης και αυτά πρέπει να συζητάμε και όχι να είμαστε στους εθέρες και να λέμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ προσωπώ την Πολωνία, μια Πολωνία που έχει κάνει ε, επιτυχώς πολλές μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουμε ακόμη πολλά πακέτα ε, για την ενέργεια που πρέπει να εφαρμόσουμε. Δεν λέω αυτά για να με λυπηθείτε, αλλά πώς συζητάμε έτσι ευρωπαϊκά ζητήματα φλού, χωρίς να λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη τις ιδιαίτερες καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Και μπορεί στα λόγια η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να ηγείται παγκοσμίω στην όλη προσπάθεια, αλλά φαίνεται να είναι και πολύ μοναχικό ηγέτη η Ευρώπη στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ και τι συμβαίνει σε άλλε χώρε του κόσμου. Βλέπουμε ε, μια μεγάλη μοναχικότητα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Η μείωση ε, των εκπομπών ρήπων λοιπόν, του διευθυντου άνθρακα ε, είναι κάτι καλό, συμφωνούμε όλοι, αλλά τελικά με αυτούς τους που πάμε, θα σώσουμε πραγματικά τον πλανήτη. Ακούστε και τα σχόλια των άλλων ε, παγκόσμιων παικτών για τη θέση της Ευρώπης. Τι είπε η Αυστραλία, τι είπε και ο Ομπάμε πριν από λίγες μέρες για αυτή τη θέση της Ευρώπης. Αυτό το παράδειγμα του εργοστασίου αλουμινίου είναι πολύ καλό παράδειγμα. Δεν παράγει πλέον στην Αγγλία, παράγει στον Καναδά. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει ε, να ακούμε με σεβασμό τις απόψεις των άλλων. Όλοι θέλουμε ένα καθαρό κόσμο και ε, ε ένα μέλλον για τον κόσμο μας. Αλλά ε, μας απασχολεί και η ενεργεία. Μιλούμε ταυτόχρονα για το νέο ε, πακέτο δημοσιονομικών προοπτικών, συζητούμε για θέματα απασχολησιμότητας. Είναι και αυτά θέματα που είναι εξίσου σημαντικά και πρέπει να συνδέσουμε τη συζήτηση ε, για το κλίμα με αυτά τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Αυτό το σύστημα backloading που προτείνει η Κομισιόν μπορεί κανείς να, να πει ότι είναι παρέμβαση στην αγορά και σε κάποιες ε, τροπολογίες επεξηγηματικές μας λέτε ότι είναι μία φορά που θα γίνει, αλλά δεν πιστεύω ότι μας πιστεύουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των σκιωδών ε, εισηγητών και σας διαβάζω τα ονόματα των άλλων που ζήτησαν το λόγο. Μήπω Μήπως ξέχασα κανέναν, η κυρία, την κυρία Γκαρδίνη. Ωραία, προτείνω να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών και να περιορίσουμε το χρόνο ε, στα δύο λεπτά, διότι αμέσως μετά έχουμε την ε, έκθεση του Πέτερ Λίζε και θα χρειαστούμε χρόνο για να τη συζητήσουμε. Ο Πέτερ Λίζε, δύο λεπτά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Διαδικαστικό. Προτείνω πάνω από δύο λεπτά για τον κάθε αγόρι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για να δίνετε μόνο δύο λεπτά. Τότε προτείνω αν συμφωνούν όλοι και ο Πέτερ Λίζε, να ε, πούμε δυόμιση λεπτά. Ο Καρλ Χάινς Φλόρενς ε, κάνει παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο και, και στην Κομισιόν θα πρέπει να δώσουμε το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Προτείνω δυόμιση λεπτά, συμφωνείτε? Ο Πέτερ Λίζε διαφωνεί. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε. Δεν θα τα είχαμε προλάβει όλα αν, συζητούσαμε, αν είχαμε να συζητήσουμε σήμερα και την ε, ε, ε, έκθεση του Ούλμερ. Θα παρακαλούσα να εφαρμόζεται από την αρχή των κανόνα περί χρόνου ομιλίας. Οι εσκιώτες εισηγητές των μικρών πολιτικών ομάδων νομίζω μπορούν να περιοριστούν και λίγο περισσότερο. Ο Ρίχαρτ Σέμπερ είναι ο υπεύθυνο συντονιστής και θα μιλήσει για τις ε, συζητήσεις εντός του και Εγώ είμαι η εισηγητής του Κοινοβουλίου για το θέμα της αποτελεσματικότητας ε, της ενέργειας ε, και το Κοινοβούλιο απέτησε την πρόταση αυτή και η αξιοπιστία μας απαιτεί να μην πούμε απλά όχι. Αν κάποιος έχει καλύτερη πρόταση να την υποβάλει, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς. Ένα όχι δεν ε, θα έδειχνε συνέπεια και μιλώ όχι μόνο στο δικό μου όνομα. Υπάρχει μια σειρά συναδέρφων από, ε, το, ε, από την πολιτική ομάδα του ΕΛΚ που πιστεύουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Λέω λοιπόν στον Μπάς Άικχαουτ ότι έχω σαφείς ε, ενδείξεις ότι ο Πέτερ στο Βερολίνο δεν, ε, δεν είναι μόνος του ε, και ότι η γερμανική θέση στο Συμβούλιο δεν θα είναι να πούμε όχι. Το πρόβλημα που έχουμε είναι τόσο μεγάλο επειδή ήδη από το 2005 είχαμε υπερβολική είχαμε κατανομή υπερβαλλικά πολλών δικαιωμάτων και ο συνάδελφος Ζωζ Μορέιρα το 2002-2013 πρότεινε ένα benchmark, ένα σημείο αναφορά. Εάν ε, το είχαμε ε, εγκρίνει αυτό και το είχαμε περάσει και στο Συμβούλιο, δεν θα είχαμε σήμερα τη συζήτηση αυτή. Αλλά παρά ήμασταν ε, γενναιόδοροι και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι και επιπλέον έχουμε και την οικονομική κρίση. Ε, και η Ρίτα Κόρχολα αναφέρθηκε στην διαδικασία μάθησης. Ε, πρέπει ε, να ξεκινάμε αργά και να μαθαίνουμε. Ε, τώρα μαθαίνουμε και δεν θα πρέπει τότε να πούμε ότι α, όχι δεν θα, κάνουμε, δεν θα μάθουμε από τα προηγούμενα και δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν η υπερβολική κατανομή από την αρχή. Οι βιομηχανίες που εκπληρούν τις προϋποθέσεις έχουν επωφεληθεί από το σύστημα ε, και θα επωφεληθούν ε, και, παρα... και περαιτέρω διότι σημαίνει ότι θα έχουν μεγαλύτερη αξία τα πιστοποιητικά που έχουν και δεν θα χρειαστούν νέα. Ε, και τέλος, πολύ σημαντική παρατήρηση και προς τον Κέλερμαν τα προβλήματα που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία έχουν να κάνουν με εθνικά μέτρα. Θα λύσουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόβλημα και μετά ε, σε εθνικό επίπεδο ε, θα ε, επιδρώνουμε την κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην έχουμε επιπλέον εθνικά μέτρα. Ε, ο Καλ Φλόρεν, Φλόρενς, ε, ναι, ο Πέτερ Λίζε με κάλυψε εν μέρη. Ε, θα πρέπει να μου εξηγήσετε γιατί για δεύτερη φορά είχαμε υπερβολική κατανομή και γιατί δεν έχουμε μάθει από τα διοικητικά μέτρα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περιορίσει την κατανομή. Νομίζω ότι η Κομισιόν δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της. δεύτερη ερώτηση προς την Κομισιόν. δεν σας αρέσει η πρόταση του συναδέλφου Γκρότε να ε, παρέμβετε μία φορά. Θέλετε δηλαδή λευκή επιταγή ώστε στο μέλλον να μπορείτε να παρεμβαίνετε κάθε έξι μήνες και όσον αφορά την τιμή των 4,80 ευρώ ή των 6 ευρώ σε ένα σημείο που βασίζεται στην αγορά, αν θέλει να το διατηρήσει κανείς, θα πρέπει να δεχτεί κανείς τις χαμηλές τιμές. Ε, η Γερμανική Τράπεζα, η Deutsche Bank και ε, τα, οι μετοχές της ε, βρίσκονται πολύ χαμηλά και οι σοφοί τις αγοράζουν. εγώ δεν τρομάζω από την χαμηλή τιμή. Μία και μοναδική παρέμβαση δεν ε, θα λύσει το πρόβλημα. Δεν ε, έχω λάβει οριστική απόφαση, αλλά ίσως η Κομισιόν ε, μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι θέλετε ένα μέσο για να παρεμβαίνετε κάθε χρόνο. Ευχαριστώ, κύριο Σκυλακάκης. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομο. Ας ξεκινήσουμε από το ETS δεν είναι ο στόχος μας, είναι το εργαλείο, το μέσο. Ε, ο στόχος μας είναι οι εκπομπές. Ποιο θέλει να εξετάζει και να θαυμάζει μόνο το εργαλείο και να μην εξετάζει το στόχο και γιατί λειτουργεί το εργαλείο. Για πρώτη φορά αγοράζουμε φτηνές ε, CDMs ε, για 0,4 ευρώ. Πριν το αγοράζαμε για 12 ευρώ σπαταλούσαμε ουσιαστικά τα χρήματα των Ευρωπαίων καταναλωτών ενέργειας. Για πρώτη φορά λοιπόν λειτουργεί πραγματικά, είναι το αντίθετο από αυτό που είπατε. Καινοτομία τώρα. Καινοτομία πού? Ε, στα φωτοβολταϊκά και στις ανεμογεννήτριες. Αυτά παράγονται στην Κίνα γιατί είναι πιο φθηνά εκεί. Έτσι έχουμε αποτύχει ε, σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής σε μεγάλο βαθμό και τώρα προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε με τρόπο όμως που δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε να ε, προωθήσουμε την ε, καινοτομία και τις επενδύσεις, συγγνώμη. Αλλά αυτοί που θα πάρουν τις επενδυτικές αποφάσεις θα έχουν τις τιμές του ETS για το, 19 και του 20 κατά νου αυτή τη τιμή εμεί θέλουμε να τη μειώσουμε, μεταφέροντας το backloading για τότε. Επομένω, για τους επενδυτές ε, είναι άσχετο. Εφόσον οι αποφάσεις για επενδύσεις σήμερα θα βασίζονται στις τιμές του 19 και του 20. Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος λοιπόν είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Κάποιοι θέλουν κρατικές ενισχύσεις και κάποιοι, κάποιες χώρες μπορούν να τις δώσουν, κάποιες άλλες όχι. Ιδίω οι χώρες του Νότου δεν μπορούν να δώσουν ενισχύσεις ε, στις, ε, στον τομέα τη ενέργειας. Επομένω, στρεβλώνουμε την ενιαία αγορά με υπόγειο τρόπο. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Γιατί κάποιοι μπορούν να δώσουν ενισχύσει, έχουν ε, πλεόνασμα ή κάτι που θυμίζει πλεόνασμα στον προπολογισμό τους. Κάποιοι εδώ ξεχνούν τους καταναλωτέ ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, στη χώρα μου έχουμε 250.000 ε, πολίτες που τρώνε από συσίτια γιατί, γιατί θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα για να πληρώσουν λογαριασμό του ηλεκτρικού. 250.000 άνθρωποι. Τους ξεχνάμε, τους λέμε θα πληρώσετε λίγο παραπάνω θα βρείτε μερικά ευρώ παραπάνω, γιατί εμεί θέλουμε να καινοτομήσουμε το 2020 κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίχαρτ Τζέμπερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ζωντανή η συζήτηση. Χαίρομαι γι' αυτό και μας δείχνει ότι με το αναδρομικό αυτομέτρο, το bank ε, loading, δεν μιλάμε για την προστασία του ε, κλίματος ε, με την ευρεία έννοια, μιλάμε για άλλα μέσα ε, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εθνικοί φόροι κλπ. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών στόχο είχε να υπάρχουν ανώτατα όρια και την εμπορία. Η βιομηχανία πληρεί ε, τις προϋποθέσεις σχετικά με τα ανώτατα όρια. Το θέμα είναι τι γίνεται με την εμπορία. Υπάρχει εμπόριο, είναι χαμηλή η τιμή. Δεν λέει πουθενά στην ε, οδηγία ότι χρειαζόμαστε υψηλή τιμή. Οι προϋποθέσεις λοιπόν που έχουμε θέσει προς την βιομηχανία ως ε, πληρούνται απόλυτα. Εάν θέλουμε κάτι άλλο πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Αλλά μπά και κρίς. Για σας ποια είναι η σωστή τιμή. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό, διότι αν έχουμε το αναδροτικό μέτρο και η τιμή ανέβει στα 6-7 ευρώ, ε, μπορεί από την επόμενη μέρα ήδη να έχουμε τη συζήτηση σχετικά με το ότι η τιμή αυτή είναι υπερβολικά χαμηλή. Τι θέλουμε λοιπόν. Όχι, να είμαστε σαφείς. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και όχι να κατηγορούμε ο ένα τον άλλον. Ε, τι θέλουμε λοιπόν, το αρχικό σύστημα λειτουργεί. Αλλά μήπω ε, δεν είναι, μήπως δεν είναι αρκετά πικρό το φάρμακο. Είμαι πεπισμένος ότι με το backloading θα πετύχουμε μόνο ανασφάλεια. Κανένας ε, δεν θα ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Και ε, είναι ωραίο το έγγραφο, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ε, θεμελιώδη μεταρρύθμιση. Και ο συνάδελφος Σκυλακάκης αναφέρθηκε στην τιμή της ενέργειας. Ε, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να μην είναι πρόβλημα αυτό, σε άλλα να είναι. Ε, το, το πρόβλημα είναι ότι πουθενά δεν λέει ότι τα χρήματα αυτά ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για καινοτόμα μέτρα. Είναι ένα τέλος που, τα, που πληρώνει η βιομηχανία για τον γενικό προϋπολογισμό. Μπορούμε να πούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για καινοτόμα μέτρα, αλλά τότε θα χρειαστούμε ε, χρόνο μέχρι το 2015 που θα υπογραφεί η Σύμβαση για το Κλίμα. Αλλά τώρα, πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σύστημα να το συμπληρώσουμε, πιστεύω ότι είναι λάθος πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελίντα Μακέβαν. Thank um, Ευχαριστώ. Ελπίζω πριν πάμε στη ψηφοφορία να το σκεφτούμε και να το δούμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, να μιλάμε και τεχνικές λεπτομέρειες και προσωπικές, αλλά μπαίνουν και θέματα ουσίας στη συζήτηση. Όσοι θεωρούν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να το σκεφτούν σοβαρά πριν ψηφίσουν. Ιδίω συνάδελφοι που στο παρελθόν υπερψήφισαν τις πολιτικές για το κλίμα και τώρα λένε όχι δεν θέλουμε προσαρμογή γιατί η αγορά έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Και όσοι, όπως και εγώ, υποστηρίζουμε την ελεύθερη αγορά, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει. Ο Ματίας τι είπε στην αρχή της συζήτηση ότι ένα από τα θέματα που τίθεται είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βρει μόνη της ε, λύσης ε, σε ό,τι αφορά τι τιμέ του άνθρακα, τα κάτι μέλη από μόνα τους αρχίζουν και παίρνουν μέτρα. Μάρτιν, το νεμόνο Βασίλειο ε, πήρε ειδικά το μέτρα για την τιμή του άνθρακα και το προσπάθησα να το ελέγξω. Η Βρετανική ήταν η τιμή που δημιούργησε το σοβαρότερο πρόβλημα. Να το δούμε, να δούμε τη διαφορά α, ανάμεσα στην αγορά τιμή του άνθρακα και τη Βρετανική τιμή. Εσύ είχε πει εκείνη τη στιγμή ότι ήταν κυβερνητική πολιτική παράλληλα που έτρεχε με τι ευρωπαϊκέ ε, παρεμβάσει. Οπότε ε, δεν είναι αυτό λυπηρό όπω συνέβη. Και είπε και ο Κρίς Ντέιβες ότι το ETS το, πρόβλημα ποιο είναι, ότι είναι συνδυασμό φαλμάτων. Το είχα πει και την πρώτη φορά. Στη δεύτερη φάση είχαμε ψηφίσει ένα κανονισμό και ε, είχαμε υπερπληθώρα πιστώσεων που πλημμύρισαν την αγορά. Άρα, όπως είπε η κυρία Κοχάλαρ, ότι δεν είμαστε παιδάκια πια. Και λέτε δηλαδή μόνο τα παιδιά μαθαίνουν στη ζωή Εσείς δηλαδή σας την και τα μάθατε όλα, έτσι. Δεν, δεν χρειάζεται να μάθετε τίποτα παραπάνω. Μα η ζωή ε, και τα δεδομένα αλλάζουν και μαθαίνουμε πάντοτε και προσαρμοζόμαστε πάντοτε. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν δεν υποστηρίξει την Κομισιόν σε αυτό το θέμα, τότε τι θα κάνετε για την κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να ερχόμαστε εδώ και να μιλάμε για μεγάλα ψηφίσματα και μεγάλα λόγια. Θα πάτε στη Βαρσοβία, στη συζητήση για το κλίμα, για να καταλήξουμε και παγκόσμια συμφωνία αν καταρρεύσει το ETS εδώ στην Ευρώπη, τι ελπίδα έχουμε να πείσουμε τους Αυστραλούς, τους Κινέζους που έχουν δικά τους συστήματα ETS και θεωρούν ότι εμείς είμαστε ένας σοβαρός εταίρος. Είστε λοιπόν πραγματικά σοβαροί εταίροι για την προστασία του κλίματος, ναι ή όχι. Πράγματι, κάποιοι ήταν πάντοτε κατά ε, της πρότασης και δεν τους ενδιέφερε σε το κλίμα. Κύριε Χαλέρη, ίσως είναι πάντοτε ακόλουθοι. Οι άλλοι όχι. Ας το σκεφτούν. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Καρτίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ήδη υπόθησαν πολλά. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση εμβάθυνσης. Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Από ό,τι άκουσα, η Ήτρε πέρας, ε, καταψηφίστηκε, συγγνώμη, ε, οριζόντια η πρόταση. Μόλις σε, μάλλον 42 άτομα υπερψήφισαν ε, την καταψήφιση της πρότασης της ε, Κομισιόν και μόλις 12 ήταν υπέρ. Α, αυτό εγώ θεωρώ δείχνει ότι δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση πρώτα απ' όλα. Και φταίει και το ίδιο το Κοινοβούλιο γι' αυτό. Και συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε σε μια τέτοια στιγμή κρίσης, τόσο βαθιάς κρίσης, να γυρίσουμε σπίτι μας και να πούμε στους ε, συμπολίτες μας ότι α, ε, και ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα αυξηθεί έτσι απλά αλλά δεν θέλω να επιμείνω μόνο σε αυτά που ήδη ακούστηκαν. Στη χώρα μου έχουμε σημαντική μείωση της παραγωγής, σε κάποιους τομείς παραγωγής φτάνουν και το 40%. Η κρίση λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοούμε όταν συζητούμε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε εναλλακτικά, δηλαδή ή πολιτική για το κλίμα ή οικονομική πολιτική πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη την βαθιά οικονομική κρίση όταν μιλάμε και για το κλίμα. Για το κλίμα είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα συνάδελφο που διαφωνεί. Από την άλλη όμω υπάρχουν και πολλές άλλε δεσμεύσει που αφορούν το πακέτο για το κλίμα, την ενέργεια, τι ανανεώσιμε, την αποτελεσματικότητα κλπ. Αλλά θέλω να σταματήσω στο εξή. Ο κ. είπε ορθά ότι υπάρχουν και οι αντισταθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για το έμεσο κόστος των ETS. Ε, τότε θα θέλαμε ένα υποχρεωτικό σύστημα, διότι αυτές οι στρεβλώσεις ε, που υπάρχουν όχι μόνο στην παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να τι μεταφέρουμε και στην εθνική μα αγορά. Από ό,τι κατάλαβα η Γερμανία και η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχουν δώσει πολύ σημαντικά ποσά προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ άλλε χώρες δεν έχουν κάνει τίποτα αυτό πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που εξαρτάται και από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρτίνη. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Από πλευρά μα θα θέλαμε μόνο να επενθυμίσουμε ότι πράγματι η Επιτροπή ξεκίνησε ε, πέρσι τον Απρίλιο ε, από την Επιτροπή υπογραμμίστηκε και τονίστηκε αυτό το πρόγραμμα. Το καλοκαίρι ε, υπήρξε μια σειρά εγγράφων που ανέλυαν την κατάσταση και σηματοδοτούσαν ε, την ε, κρισιμότητα της κατάστασης, δηλαδή της υπερπληθώρας προσφοράς που έχουμε στην Ευρώπη, γιατί κάτι πρέπει να γίνει με πιο λογική κατανομή της προσφοράς χωρί να επηρεάζεται η οροφή που έχει τεθεί. Πριν από τρει μήνε, κατόπιν αιτήματο των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ε, κατέθεσε συγκεκριμένε προτάσει, όχι μόνο για την διασπορά με, και κατανομή με καλύτερο τρόπο και πιο λογικό τρόπο αυτών των ε, δικαιωμάτων, το λεγόμενο bank loading που θα περάσει από την Επιτροπολογία, αλλά και μια έκθεση ε, για την αγορά που θα αναλύει περαιτέρω την κατάσταση και θα κάνει προτάσει για διαφορετικά μέτρα. Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τα Διαθετικά αυτά μέτρα. Πριν από τρει μήνε είχαμε μια τιμή 8 ευρώ όταν έγινε η πρόταση. Πέρασε ο καιρό για να συζητηθεί και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο η πρόταση και η τιμή έχει πέσει κι άλλο. Το προηγούμενο εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ακυρώθηκε μία από τι δημοπρασίε, αναφέρθηκε προηγουμένω, και αυτό είναι ένα σύμπτωμα αυτή τη υπερπροσφορά. Μπορούμε λοιπόν με λογικό τρόπο να το δούμε αυτό και να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί και θα συνεχίσει να παίζει να πέφτει συγγνώμη, η τιμή, ε, το οποίο επιβεβαιώνουν και όλοι οι αναλυτές. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Πριν από αυτό όμω πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και κάτι για να σώσουμε και να συζητήσουμε. Αναφέρθηκε ότι ήδη κάποια κράτη-μέλη έχουν λάβει εθνικά μέτρα και είναι πολύ πιθανόν και μεγάλο κίνδυνο. αν πέσει κι άλλο η τιμή ήδη σήμερα να ε, θεσμοθετηθούν νέα μέτρα. Και αυτό είναι κατακαιρματισμό της εσωτερική αγοράς ε, που είναι πολύ σημαντική για την βιομηχανία. Στη διαδικασία διαβούλευση, ουσιαστικά όλη η βιομηχανία είπε ότι στηρίζει το ETS, στηρίζει τις ε, ε, αναδιαρθρώσεις, όμως αν δεν ακολουθήσουμε αυτή την πιο λογική προσέγγιση για καλύτερη κατανομή και ε, τότε αυτή η στήριξη δεν είναι προφανής. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω ότι πράγματι σε διεθνέ επίπεδο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην εμπορία ρήπων, εκπομπών. Βλέπουμε ε, τι συμβαίνει και στην Αυστραλία και στην Κίνα και εξελίσσεται ραγδαία κατάσταση. Η Ευρώπη δεν πήγε αρκετά γρήγορα, ε, αναφέρθηκε. Ε, ήδη στη δεκαετία του 1990 είχαμε μακροσκελήσεις συζητήσεις ε, για άλλες πολιτικές όπως ο φόρος ε, άνθρακα που τελικά δεν ε, καρποφόρησε και έτσι είναι φυσιολογικό και άλλες ε, χώρες να χρειάζονται χρόνο πριν καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα. Είναι όμως πολύ καλή εξέλιξη για παράδειγμα το ότι συμβαίνει στην Κίνα και ότι ήδη μας έχουν πει, έχουν συγκρίνει τις διάφορες ενέργειες και έχουν επιλέξει το δικό μας σύστημα, το ETS, όσο πιο αποδοτικό και λειτουργικό. Και παρακολουθούν και βλέπουν ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας έχουν ε, αντιλήσει πολύ ε, δυνατά και σημαντικά ε, μηνύματα από την συμφωνία του 2008, τα οποία μόλις τώρα θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Ξεκινήσαμε την τρίτη φάση το 2013. Επομένω, βλέπουμε ότι πράγματι ε, μαθαίνουμε από την εμπειρία μας και προσαρμόζουμε και την προσέγγιση μα. Τέλο να πω ότι πράγματι για τα διευθυντικά μέτρα συζητούμε με τα ενδιαφέρομενα μέρη και ε, υπάρχει τέτοια διαβούλευση. Θα υπάρξει και συγκεκριμένη συνεδρίαση με τα ενδιαφέρομενα μέρη, του stakeholders. Επομένω, είναι ένα στοιχείο που πάντα ε, είναι, έχουμε κατά νου. Τέλο, για το blind check. Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχύει ότι η Επιτροπή θέλει να έχει την ε, έσχατη εξουσία να παρεμβαίνει ε, στην αγορά. Υπάρχουν και διατάξεις στη συνθήκη. Ε, η Επιτροπή έχει την ευθύνη και υποχρέωση να δίνει αξιολόγηση αντικτύπου, κάτι που έχουμε πράξει, για να παρεμβαίνει όταν υπάρχει στήριξη και από το κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο. Επομένως, αυτό που αναφέρθηκε δεν αληθεύει, ποτέ δεν θα συμβεί. Ε, αυτή η κατάσταση ισχύει μόνο τώρα, είναι μια ακραία κατάσταση και δεν πιστεύουμε ότι θα ισχύει ε, συχνά. Όμως έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα πρέπει να ενεργήσουμε. Αυτή ήταν η τελευταία έκκληση της Κομισιόν. Έχουμε σημειώσει τις παρατηρήσεις σας, ακούσαμε τις επιφυλάξεις σας ιδιαίτερα εδώ από τα δεξιά. και ουσιαστικά δεν ε, υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο πρόβλημα. Δεν ε, διαφωνώ με αυτό. Μόνο χρόνο κερδίζουμε με την πρόταση αυτή, ε, αλλάζοντας το χρονοδιάγραμμα. Δεν μιλάμε για τίποτα παραπάνω. Ε, ούτε και εγώ θεωρώ ότι ψηφίζουμε επί της ουσίας του συστήματος εμπορίας ε, εκπομπών. Καταλαβαίνω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, άκουσα αυτά που είπε ο Έλληνας συνάδελφος ο κύριος Κυλακάκης. Άκουσα και αυτό που είπε ο Μάρτιν Κάλαναν που μίλησε για ε, τη δική του εκλογική περιφέρεια. Ξέρουμε και άλλα παραδείγματα, αλλά Όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, το πρόβλημα υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Και όσον αφορά την, ε, τις αποζημιώσεις. Ε, άκουσα πρόσφατα για κάποιον ε, πάροχο υπηρεσιών που θεωρήθηκε ότι παρέχει υπηρεσίες Φιλικέ προς το περιβάλλον και γι' αυτό ε, έχει ε, κερδίσει ένα πλεονέκτημα απέναντι στου ανταγωνιστές του. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο πραγματικά ε, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, διότι νομίζω σαφές είναι ότι κανείς εδώ δεν θέλει να μεταφερθούν θέσεις εργασίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά κάποιος που θέλει μια βιώσιμη οικονομία χρειάζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μια καλή ε, βιομηχανία ε, ε, ατσαλιού στην Ευρώπη και άλλα. Μπορώ να σας πω τι είδαμε στην Τόχα σε συζητήσεις ε, με ε, Βραζιλιάνους και Ιαπωνέζους και άλλους. Θα υπάρξει ένα σύστημα. Ε, έχουμε στην ημερήσια διάταξη και την έκθεση του Πέτερ Λίζε. Θα γίνει σαφές ότι στις διεθνείς αερομεταφορές θα ανοίξουμε ε, την πόρτα για άλλους τομείς επίσης για να έχουμε σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών. Ε, τι βλέπουμε στον κόσμο. Βλέπουμε τώρα φόρο επί των αερομεταφορών και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 50% των εσόδων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για μέτρα προσαρμογής και για την προστασία ε, του κλίματος. Ε, δεν ε, είναι στη διάθεση των Υπουργών Οικονομικών τα χρήματα αυτά. Ίσως θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι το πρόγραμμα αυτό δεν ε, έχει στόχο την ε, αναχρηματοδότηση των ε, εθνικών προϋπολογισμών. Πρέπει να χρηματοδοτηθούμε τα χρήματα αυτά μέτρα προστασίας κατά της αλλαγής του κλίματος. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να στείλουμε σαφή μηνύματα. Πρέπει να δείξουμε ότι το σύστημα λειτουργεί πράγματι λειτουργεί. Δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα είχε με μια συγκεκριμένη τιμή. Το είπε αυτό η κυρία Κορόλα, το είπαν και άλλοι. Είχαμε ε, τη συναδελφό Εύριν από το ΕΛΚ ε, και Ε, είχε μιλήσει για κατώτατες ε, ε, τιμές, αλλά πολλοί φοβήθηκαν ότι οι τιμές θα εκτοξευθούν. Το θέμα λοιπόν είναι μήπως στο μέλλον χρειαζόμαστε βαλβίδα ασφαλείας και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Υπάρχουν και άλλους τομείς όπου ε, δεν έχουμε ε, ανώτατες και κατώτατες ε, τιμές όπως στην Γεωργία. Εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό. Θα πρέπει να βελτιωθεί. Και Από όλα όσα άκουσα σήμερα θα προσπαθήσω να τετραγωνίσω τον κύκλο, να ε, ε, μοιράσω μια συμβιβαστική πρόταση που να καλύπτει πολλούς. Πρέπει να υπερασπιστώ τη θέση του Κοινοβουλίου, διότι ζητήσαμε από την Κομισιόν να υποβάλει σχετική πρόταση. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά, τον αριθμό των πιστοποιητικών, ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλειοψηφία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αξιόπιστο που να μην δημιουργεί περισσότερη ανασφάλεια στον τομέα αυτόν. Αυτό είναι σαφές. Όταν λοιπόν διατυπώσω την συμβαστική μου πρόταση, παρακαλώ να την υπερψηφίσετε θα έχω και σχετικές συζητήσεις ε, με τις διάφορες ε, πλευρές αλλά παρακαλώ να μην ε, απορρίψουμε την, απλά την πρόταση αυτή αλλά με ευρία πλειοψηφία να λάβουμε απόφαση και να δείξουμε και στον έξω κόσμο ότι μπορούμε να βρούμε εδώ συμβιβασμούς. το σύστημα αυτό τώρα στην 20η ε, επέτειο της εσωτερικής αγοράς ε, είναι καλό. Κάποια προβλήματα δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο με διάφορους φόρους και δεν έχω καμία διάθεση ε, να έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα εθνικής φορολογίας όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγουμε την ευρωπαϊκή οδό, επιδιώκουμε τον συμβιβασμό, ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα εμπορίας εκπομπών. Στην Επιτροπή μας ε, θα ψηφίσουμε στις 19 Φεβρουαρίου και δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία για την Ολομέλεια. Το Συμβούλιο καλείται να κινηθεί, ώστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα και με το Συμβούλιο, διότι έχει να κάνει με το κεντρικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του κλίματος, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή και τώρα δίνω το λόγο στον επόμενο εισηγητή, τον Πέτερ Λίζε, που θα μας ε, μιλήσει για την πρόταση Stop the Clock ε, της Κομισιόν. Ε, μήπως ε, να περιμένουμε δύο λεπτά. Ε, ώστε να καταλήψουν την αίθουσα όσοι θέλουν. Ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους επισκέπτες μας που δεν υπήρχαν αρκετές θέσεις για να καθίσετε. Αυτό ε, ήταν ε, μια παράβλεψη της διοίκησης εδώ. Ο Πέτερ Λίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Οι δύο εκθέσεις αυτές συνδέονται στενά μεταξύ τους. και οι δύο έχουν να κάνουν με την εμπορία εκπομπών. Και οι δύο έχουν να κάνουν με το αν πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική του κλίματος, αν είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε την ε, οδό που ήδη έχουμε ανοίξει ή μήπως απλά θέλουμε να μην κάνουμε τίποτα. Ε, επειδή θεωρούμε ότι η πολιτική του κλίματος έχει αποτύχει. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο την ε, πολιτική για την αλλαγή του κλίματος ε, και ε, να κοιτάμε και τι γίνεται εκτός Ευρώπης. Αλλά η παρέτηση δεν είναι καλή στάση, ούτε θα κάνει πιο αξιοπιστή την Δύο λόγια για την γνωμοδότηση της Ήτρε. Πιστεύω ότι η τιμή θα πέσει περισσότερο. Και υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε περισσότερα εθνικά μέτρα πρόκειται ίσως για μια πύριο νίκη. και αν έχουμε τέτοια εθνικά μέτρα δεν ε, πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα. Όσον αφορά τις αερομεταφορές, έχουμε εδώ να κάνουμε με μια άλλη ε, σημαντική επιτροπή του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Μεταφορών και μας πιέζει ο χρόνος. Ε, θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση αυτή ε, και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο συνάδελφος ε, ε, είναι παρόν και επανειλημμένα είχαμε συνεννοήσει για να βεβαιωθούμε ότι οι δύο επιτροπές δουλεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ λοιπόν τον Ματιό Γκρός καθώς και τον πρόεδρο Brian Simpson. Ε, στο Συμβούλιο Ομόφωνα και στο Κοινοβούλιο με 90% πλειοψηφία ε, υπερψηφίστηκε η πρόταση, ε, διότι έχουμε δει να διπλασιάζονται οι εκπομπές στον τομέα των αερομεταφορών από το 1990 και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για δράση. Η πρότασή μας είναι μάλλον μετριοπαθής, δεν μιλάμε για πλήρη ε, πληστηριασμό ε, και η ανώτατη τιμή δεν είναι 15-20%, είναι 5%. Ε, η επιβάρυνση για τους καταναλωτές δεν είναι πολύ μεγάλη. Στη Ryanair είναι 25 cents, 25 λεπτά ανά πτήση. Ο αναπληρωτής πρόεδρος μας, ε, Κερπράντη, έχει δραματοποιήσει πολύ τα πράγματα. Ε, ακόμα και για πτήση από το Χίθρο στην Κίνα στοιχίζει λιγότερο από ένα καφέ στο αεροδρόμιο ε, το, η επιπλέον επιβάρυνση. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να δραματοποιούμε τα πράγματα. Ε, για την Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και την Επιτροπή Μεταφορών είναι σαφές ότι θα πρέπει τις ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις διπυρωτικές αιτήσει ε, που ξεκινούν από την Ευρώπη. Ε, διότι τα δύο τρίτα των εκπομπών συνδέονται με υπερπόντιες πτήσεις. Και έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. πολλές τρίτες χώρες είναι επικριτικές απέναντι στο σύστημά μας. Έτσι ήταν τότε που το συστήσαμε, αλλά τουλάχιστον από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, είχαμε λάβει κάποια σήματα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ε, πήγα λοιπόν στην Ουάσιγκτον και είχα συνομιλίες και ε, το γενικό μήνυμα ήταν περιμένετε να φύγει ο Μπούς, είτε έχουμε τον Ομπάμα είτε έχουμε τον Μακέιν, θα αλλάξει η, πολιτική, ε, η κλιματική πολιτική των ΗΠΑ. Αλλά έχουμε απογοητευτεί διότι οι Αμερικανοί είναι οι ε, σημαντικότεροι αντίπαλοι μας εδώ πέρα. Ο Ομπάμα έχει πάρει Νόμπελ ε, ειρήνης, αλλά μήπως θα πρέπει να του πάρουν πάλι το βραβείο διότι ο Ομπάμα βρίσκεται στην αιχμή των αντιθέσεων. Ο ο Τζον Κάρι, αρμόδιος ε, υπουργός, έχει υποβάλει σχετική πρόταση. Εάν ε, θέλει να έχει κάποια αξιοπιστία θα πρέπει να αλλάξει τη θέση των Γερμανών στο θέμα αυτό. Ε, νομικά δεν στηρίζεται η ε, απόρριψη της πρότασης. Ε, το ΔΕΚ την έχει εξετάσει αναλυτικά και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο η πρότασή μας αυτή. Στην αιτιολογική έκθεση σας έχω κάποια σχέδια. Τα εθνικά μέτρα περνούν καλύτερα κατά κάποιο τρόπο. Δεν επικρίνονται τόσο πολύ εσωτερικά, ε, νομικά δεν αμφισβητούνται ούτε σε διεθνές επίπεδο. Ε, το αποτέλεσμα ε, του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας, της Γερμανίας είναι πολύ, οι φόροι αυτοί είναι πολύ ψηλότεροι από ε, το ETS και δεν υπήρχαν ε, δράσεις ε, διεθνών αερογραμμών κατά παρότι η Air France πρέπει να πληρώσει τον Αμερικανικό φόρο γενικά παρότι ξένες αερογραμμές πρέπει να πληρώσουν το φόρο αυτό στις διάφορες χώρες. Τα εθνικά μέτρα αποτελούν πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση ωστόσο γίνονται αποδεκτά χωρίς επικρίσεις. Ε, σας έχω μοιράσει και έναν πίνακα όπου ε, φαίνονται ε, οι επιβαρύνσεις από τα εθνικά μέτρα που είναι πολύ ψηλότερες. Οι αερομεταφερές είναι διεθνής δραστηριότητα, η προστασία του κλίματος είναι διεθνές συμφέρον. Όσοι λοιπόν συμμετείχαν στις αντιδράσεις στα θεσμικά όργανα Ε, σε αυτούς ε, θέλουμε να πούμε, ε, είχαμε ήδη πει τότε ότι αυτό που θέλουμε είναι μια, εθνική, μια διεθνής συμφωνία. Αλλά στην Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας δεν είχαμε δει να υπάρχει βούληση για κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως ελπίδα στις 9 Νοεμβρίου του 2012 Ε, ε, συνεδρίασε το Συμβούλιο της Ενσόργανος Πολιτικής Αεροπορίας ε, και αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2013 να βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει λύση ακόμα, αλλά αυτοί που γνωρίζουν καλά τα θέματα αυτά λένε ότι υπάρχει η ελπίδα και μάλιστα ε, ε, η ηγεσία, η διεύθυνση της, της Διεθνής Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ε, επιδεικνύει επαρκή βούληση, ίσως όχι απαραίτητα τα κράτη-μέλη. Ε, γι' αυτό έχουμε και εμείς την πρόταση αυτή Stop the Clock. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας να στείλει ένα θετικό μήνυμα προς τους εταίρους και η πρόταση προβλέπει οι διπηρετικές πτήσεις που ξεκινούν από την Ευρώπη ή καταλήγουν στην Ευρώπη να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ε, θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου να παραδώσουν τα πιστοποιητικά του ε, και να πληρώσουν τα ενδεχόμενα δικαιώματα ανάλογα με την ενεργειακή αποδοσή των ε, αεροσκαφών ε, και αυτό μάλιστα για ένα χρόνο. Τα ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκέ πτήσει θα παραμείνουν εντό του συστήματο και ακόμα και αν πραγματοποιούνται από αμερικανικές ή κινέζικες αεροπορικές εταιρείες. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή που εδρεύει η εταιρεία, αλλά η πτήση που πραγματοποιείται. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε γρήγορα την πρόταση αυτή, διότι στις 30 ε, Απριλίου έχουμε την ε, ε, καταληκτική ημερομηνία και αν καθυστερήσουμε η Κομισιόν δεν θα το εφαρμόσει αυτό. Είμαστε όμως συνομοθέτες και αν δεν αλλάξουμε κάτι θα πρέπει η Κομισιόν να εφαρμόσει την παλιά νομοθεσία. Ε, δηλαδή ή θα περάσουμε την πρόταση αυτή ή θα εφαρμόσει η Κομισιόν την παλιά νομοθεσία χωρίς τροποποίηση. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε γρήγορα μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών. Οι προτάσεις τροπολογίας μου δεν είναι ε, ουσιαστικά τροπολογίες, είναι διευκρινήσεις ε, μάλλον της ε, πρότασης της Κομισιόν. Πρόκειται για μικρές βελτιώσεις στο κείμενο, δεν πρόκειται για κάποια σημαντική τροποποίηση. το μόνο που θα θέλαμε είναι, εάν δεν γίνει τίποτα στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας το Σεπτέμβριο, και εάν δεν υπάρξουν πραγματικά βήματα πρόοδου, τότε να μην παραιτηθούμε, αλλά να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον νόμο. Δεν μπορούμε 10 χρόνια να μην κάνουμε τίποτα άλλο, ο χρόνος περνάει, το ρολόι τρέχει. Καθιστούμε σαφέ λοιπόν ότι θα γίνει ε, αυτό ε, αν δεν περάσουμε την πρόταση. Ε, καθιστούμε επίση σαφέ τι περιμένουμε από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου σε λίγου μήνε. Πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία που καλύπτει όλου. Απλά θα πρέπει να είναι σαφέ τι θα γίνει στο μεταξύ. Εάν, για παράδειγμα, σε πέντε χρόνια τεθεί σε ισχύ μια διεθνής συμφωνία ε, μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε το σύστημά μας. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα, αλλά δεν ε, θα πρέπει να ε, αμφισβητήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτή είναι η βούληση όλων των εμπειρογνωμόνων με τους οποίους είχα επαφή από τους από διάφορες επαγγελματικούς κλάδους, από τα κράτη-μέλη κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πέτερ Λίζε. Είμαι ε, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ως όδης εισηγητής και είχα εργαστεί πάνω στην αρχική έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Το ανέφερα αυτό και στην προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε μια διεθνή συμφωνία για, την, ε, για τις αερομεταφορές, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είμαστε ικανοί να συμφωνήσουμε σε ένα συμβιβασμό και στην ε, πρόταση αυτή με την οποία σταματάμε το ρολόι όσον αφορά τις ε, εξωευρωπαϊκές ε, πτήσεις μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Έγινε σαφές αυτό απέναντι στις ε, αντιπροσωπείες ε, του Κοινοβουλίου που στάλησαν στην Τόχα κατά τις ε, συζητήσεις μας με τους Κινέζους και άλλους που σημείωσαν τις θέσεις μας και θεωρούμε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με αυτά που προτείνει ο εισηγητής. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα χρονικά περιορισμένο μέτρο που βασίζεται στους υφιστάμενους μηχανισμούς όσον αφορά την τιμή. Ε, η εκλογική μου περιφέρεια βρίσκεται στην βορειοδυτική Γερμανία, όπως συμπεριλαμβάνονται όλα τα νησιά και πληρώνω πιο πολλά για ε, μία πτήση 50 χιλιόμετρων ε, από ότι για μία πτήση από τη Φραγκφούρτη ε, στη Washington ε, και πρόκειται για μικρό αεροπλάνο. Ε, δεν υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις απέναντι στα εθνικά μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι το ότι οι πτήσει ε, θα πρέπει να εμπίπτουν στο σύστημα ε, εμπορία εκπομπών, διότι είναι διεθνή δραστηριότητα ε, και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε εάν εξετάσουμε τους φόρους στις διάφορες χώρες είναι ε, μπορεί να σηκωθεί τρίχα ε, ε, κάποιου και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε σαφώς ότι δεν είναι αυτή η οδός που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Όταν ο καταναλωτής θέλει να πάει διακοπές με αεροπλάνο, θα πρέπει να συνδέεται η τιμή του, της πτήσης και με την προστασία του κλίματος και θα δεν θα πρέπει να κλείσουμε την πόρτα σε διεθνές επίπεδο, αλλά να επιδιώξουμε μια διεθνή συμφωνία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την πρόταση της Κομισιόν. Σίγουρα θα συζητήσουμε μεταξύ μας οι σκιώδεις Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία πρόταση τροποποίησης θα ήθελα λοιπόν να περιοριστώ σε αυτά. Ο συνάδελφος Chris Davis από τους Φιλελεύθερους, παρακαλώ. Thank you, Chairman. So we continue to discuss... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άρα συνεχίζουμε να συζητάμε το σύστημα ETS. Συζητήσαμε πριν το backloading. Η Ήτρε απέριψε την πρόταση και η τιμή του άνθρακα κατέρευσε στα 2,8 ευρώ ήδη. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πως μέχρι το τέλος της ημέρας δεν έχουμε καθόλου πολιτική για το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το τι Βλέπω την πρόταση η οποία ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση κομισιών. Τι θέλουμε. Θέλουμε μια διεθνή συμφωνία. Προσπαθούμε να ασκήσουμε μια πίεση από ευρωπαϊκής πλευράς με ένα νομοθετικό κείμενο. Έχουμε κάθε δικαίωμα. Η Κομισιόν εδώ πολύ απλά χρησιμοποιεί την νομοθεσία αυτή ως ε, μέσο για να κερδίσει χρόνο ώστε να προσπαθήσει να διασφαλίσει μια διεθνή συμφωνία. Και αυτό το τελικό αποτέλεσμα για όλους μας, πιστεύω, το, το επιθυμητό για το Κιώτο. Α, βλέπω ότι διαφοροποιούμε όλο και περισσότερο τις ευθύνες μας, αυτό κάνουμε αλλά να μια ευκαιρία που μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Μπορεί σε λίγου μήνες αυτό να εξατμιστεί, να μην καταλήξουμε σε κάτι ουσιαστικό. Δεν ξέρω. Θα δούμε τότε τι θα κάνουμε. Θα είναι δύσκολη κατάσταση. Να επιταχύνουμε και να διακινδυνεύσουμε μία επιθετική άτσαλη απάντηση των Κινέζων ή ακόμα και έναν εμπορικό πόλεμο. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να διαπραγματευτούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Πάιχαουτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Κρίς, Καλό είναι να πω και εγώ ότι όταν βλέπουμε να καταραίουν όλο και περισσότερο οι τιμές του άνθρακα είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να μην κατανοούν ε, τη σοβαρότητα του θέματος. Δηλαδή δεν ξέρω πού πρέπει να φτάσουν οι τιμέ για να πιστούμε. Να... Ίσως κάποια να κοβιστεί αν η τιμή του άνθρακα φτάσει στο μηδέν. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι πόσο σοβαρά παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ε, πολιτικής για το κλίμα. Αυτό που εκπλήσει σε έναν βαθμό είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ευρώπη με επιτυχία κατάφερε να ξεκινήσει μία συζήτηση α, σε παγκόσμιο επίπεδο για να κάνουμε κάτι για την ε, πολιτική α, αεροπορία. Η συζήτηση ξεκίνησε με το αλλά τελικά σταμάτησε. Οπότε τώρα τα πράγματα δεν ξέρουμε προσωπικά κάτι τι κινούνται. Είναι θολό το τοπίο. Τώρα πώς λοιπόν η Κομισιόν θα αλλάξει και θα πει σταματάμε το ρολόι. Μα το ρολόι έχει ξεκινήσει να χτυπά. Γιατί να σταματήσει. Τώρα είμαστε ήδη μέσα στο πρόβλημα και ελπίζουμε ότι η ΚΑΟ θα κάνει κάτι. Και αν δεν κάνει κάτι, πώς μετά θα ξαναβάλουμε σε λειτουργία το ρολόι. Αν δούμε και τη διάθεση του Συμβουλίου και του Νομβουλίου, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι θα ξαναβάλουμε μπροστά το ρολόι. Δηλαδή, άρχισε κάτι να λειτουργεί και το σταματήσαμε, γιατί φοβόμαστε ποια είναι η άποψη κάποιων άλλων παγκόσμιων εταίρων, αλλάξαμε τη στρατηγική μα και χωθήκαμε μόνοι μα στη γωνία. Και είναι δύσκολο να βγούμε από αυτή τη θέση. Και αν ο ΙΚΑΟ δεν τα καταφέρει, θα ξανακάνουμε τη συζήτηση. Να ξαναρχίσει το ρολόι να χτυπάει ή όχι. Ε, ήδη ε, έχουμε τη στάση του χαμένου, του ιτημένου. Δεν κατανοώ γιατί αλλάξαμε στρατηγική ενώ δούλευε. Έπρεπε να συνεχίσουμε την πίεση προς τις χώρες. Απλά Εμεί υποχωρήσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από την Κομισιόν. Αν ο Ικάο δεν κάνει τίποτα, δεν τα καταφέρει, πώς θα ξαναρχίσει να χτυπάει το ρολόι. Θα ήθελα να ακούσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί απλά δεν κατανοώ αυτή τη νέα στρατηγική. Επίσης, αν μπορώ να αναφερθώ και πάλι για μία φορά στην αεροπλοεία. Η αεροπλοεία δεν καταβάλει ΦΠΑ δεν πληρώνει ε, φόρους καυσίμων όπως όλοι μας. Οι κρατικές ενισχύσεις προς είναι πολύ μικρές. Εμείς επιδοτούμε τις αεροπορικές εταιρείες, επιδοτούμε την πολιτική αεροπορία παντού. Και να, μια ευκαιρία κάτι να πληρώσει, κάτι να έρθει να ε, πληρώσουν τις και για αεροπορία η πολιτική και λέμε «Α, τελικά δεν συμφωνούν, οπότε σταματάμε το ρολόι». Μα τι κάνουμε τελικά στην Ευρώπη. Λένε κάποιοι ότι κλείνουν επιχειρήσει λόγω τη πολιτική μα για το κλίμα. Ε, αυτό δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ξυπνήστε. Δεν νιώθω καμία ανάγκη να υποστηρίξω αυτή την πρόταση να σταματήσει το ρολόι. Ε, θέλω να με πείσει η Κομισιόν με πιστικά επιχειρήματα. Και κλείνοντα να πω ότι σε μία από τις τροπολογίες μας λέμε ότι θέλουμε να είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, ποια έσοδα τέλο πάντων, α ελπίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, στο θεωρητικό επίπεδο, να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα για την διεθνή χρηματοδότηση των πολιτικών για το κλίμα. Αν βλέπουμε τις τιμές να πέφτουν τόσο δραματικά, ακόμα και αυτές οι τροπολογίες είναι μόνο θεωρητικού χαρακτήρα και είναι τελείως περιττές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chairman. Um, I... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, να απαντήσω συντομία στην ε, ερώτηση του Μπάς, γιατί προτείνει τώρα η Επιτροπή, είναι ότι ε, επέμεναν πάρα πολύ, ήταν απόλυτο ότι όχι, δεν πρόκειται να το προτείνουμε αυτό, δεν πρόκειται να ενεργήσουμε, ε, μέχρι τη στιγμή που οι Κινέζοι απειλήσαν ότι θα σταματήσουν να αγοράζουν αεροσκάφη της Airbus. Αυτό έγινε λοιπόν. Ό,τι και λέει η Επιτροπή, ξέρουμε ότι αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα πίσω από την απόφαση. Όπως και να έχει, ε, την αποδεχόμαστε, ε, θα τη στηρίξουμε και για την έκθεση του κυρίου Λίσε. Και κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα δόκιμο ότι αν ε, προχωρήσουμε με αυτές τις εμειώσεις πρέπει να γίνουν παγκοσμίω και διεθνώς. Αν αυτό βοηθήσει να αναλυφθεί δράση στον ΙΚΑΟ, τότε αυτό είναι καλό. Θα δούμε τι θα γίνει για εκεί τον επόμενο Σεπτέμβριο. Βεβαίω και υπάρχει πολιτική πίεση τώρα σε αυτούς ε, να υπάρξει σφαιρική και γενική συμφωνία. Γιατί ξέρουμε ότι οι οραγραμμέ έχουν την κακή ε, συνήθεια να κάνουν διεθνή ταξίδια και να φεύγουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές. Ε, και η φορολόγησή του θα πρέπει να γίνεται σε διεθνή παγκόσμια βάση. Αυτό είναι και πολιτική και γεωγραφική πραγματικότητα και ελπίζω να υπάρξει συμφωνία στον ΙΚΑΟ Εν τω μεταξύ, η πρόταση αυτή είναι λογικό να τύχει στήριξη και εμεί θα τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ, Μάρτιν. Ευχαριστώ τον Μάρτιν Κάλεναν και ο συνάδελφος Σιμάνσκι, παρακαλώ. Δεν είναι παρόν. Ματιό Γκρός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών. Ε, είχαμε ήδη εκεί συζήτηση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να φτάσω στα ε, συμπεράσματα που, στα οποία καταλήξαμε εκεί πέρα. Ελπίζουμε ότι η ΚΑΟ κάτι θα κάνει τελικά. Όλες οι πολιτικές ομάδες γενικά στηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν. Ωστόσο, τονίζουν ότι αυτή η εξαίρεση, αυτό, αυτή η παρέκκληση stop the clock θα ισχύει για ένα χρόνο. Δεν ε, θέλουμε να ανοίξουμε άλλες ε, συζητήσεις. Ε, μένουμε στις θέσεις μας. Και μετά τη συνέλευση ΚΑΟ φέτος ελπίζουμε ότι τελικά θα σημειωθεί η πρόοδος. Και δεν θα θέλαμε να βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων, όπως έγινε το 2004 χωρίς συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Ε, τελευταία παρατήρηση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διμερείς ε, συμφωνίες που έχουμε με διάφορες περιφέρειες. Ίσως θα πρέπει να ε, προσέξουμε περισσότερο τι υπάρχει από πλευράς νομοθεσίας. Υπάρχει το Open Sky στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, ε, ίσως σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, αν το λάβουμε αυτά υπόψη μας, να είναι πιο εύκολος ο ρόλος μας και Ε, να προλάβουμε επικρίσεις. Ε, έτσι νομίζω θα μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς και αυστηροί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Ο Φόλκερ Κράμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, όταν ανακοινώθηκε πέρσι η ευνηδιαστική ε, πρόταση της Κομισιόν, είχα μια συζήτηση με τον ε, Πέτερ Λίζε. Έκανα τότε την πρόταση δεν, ότι δεν, έχει τόσο πολύ νόημα να φορτώσουμε αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές αερογραμμές το, το πρόβλημα. Παρακαλώ λοιπόν να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το θέμα των ε, τρίτων ε, χωρών, ε, αλλά να σκεφτούμε και λίγο τι πετυχαίνουμε αν έχουμε ένα αποκλειστικά ευρωπαϊκό σύστημα. Το κλίμα δεν θα επωφεληθεί πάρα πολύ. Να λάβουμε υπόψη μας γενικά τη θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες, η οποία δεν είναι πολύ καλή. Και ε, αν επιβάλλουμε κάτι αποκλειστικά στις ε, ε, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, μάλλον δημιουργούμε πρόβλημα και δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε να αλλάξουν θέση. Η αλλαγή του Υπουργού δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα. Ο Ομπάμα έχει απαγορεύσει ε, αμερικανικές εταιρείες να ε, συμμετέχουν στο, σύστημα, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Η γραμμή λοιπόν του Μπούς και του Ομπάμα είναι η ίδια, ε, όπως επίσης και η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και βέβαια δεν απομένει στην Κομισιόν άλλη λύση από το να υποβάλει την πρόταση αυτή. Έχουμε μέχρι στιγμής αγνοήσει τις αντιθέσεις ε, των ε, τρίτων ε, χωρών και τις έχουμε υποτιμήσει. Αναφέρθηκε ο Μάρτιν Κάλαναν σε αυτό. Οι τρίτες χώρες απειλήσαν με αντιμέτρα, αλλά αυτό δεν ήταν μπλόφα. Ήδη έχουμε δει κάποια ε, πρώτα βήματα ε, αντίστοιχων μέτρων από άλλες χώρες. Δεν ε, θα πρέπει λοιπόν να διακινδυνεύσουμε σε ένα χρόνο να μην έχουμε πια καμιά επιλογή άσχετα από το τι θα γίνει στην ΙΚΑΟ. Και μία τελευταία παρατήρηση για τις δαπάνες. Οι αντιρρήσεις των τρίτων χωρών δεν είχαν να κάνουν με τις δαπάνες του ε, συστήματος. το θέμα είναι ότι οι τρίτες χώρες δεν θέλουν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικό τους εναέριο χώρο. Ε, σε αυτό το επιχείρημα δεν έχει απαντήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε ο Πετελίζε στην εκθεσή του. Εάν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε, εάν θέλουμε ε, να έχουμε οποιοδήποτε μέσο ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κυβερνά τον κόσμο. Δεν αποφασίζουμε εμείς το παιχνίδι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς και Ε, τελικά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε καταλήξει το αργότερο μεταδικό ότι ε, δεν ε, έχουμε εμείς η ηγετική θέση στον κόσμο, δεν αποφασίζουμε εμείς. Η κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ. Θα επιστρέψω, αν θέλετε, στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε σήμερα το πρωί, στην οποία συμμετείχα. Υπήρξε μια ε, τροπολογία απόρριψη ε, που υπερψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πρέπει να απογραμμίσω. Βεβαίω, δεν ε, συμφωνήσαμε καθόλου με την θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτου λεχθέντω, για την έκθεση Λίζε, συμφωνώ με τις τελευταίες παρεμβάσεις και να πω σε ορισμένους συναδέλφους ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αφελείς. αν δεν υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας και αν δεν εφαρμόζεται, τότε ε, κάνουμε λάθος. Και βεβαίως υπάρχουν και ε, ορισμένα μέτρα με συγκεκριμένες ε, απειλές και εκβιασμούς από πλευράς ακίνας που ε, αφορούσαν και την, ε, την ε, πώληση αεροσκαφών της Airbus. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με του συναδέλφου που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφασίσει ε, τι σημαίνει σε όλο τον κόσμο. Α ελπίσουμε ότι κάποια μέρα θα υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών, όμω μέχρι τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έτσι στηρίζω τον συνάδελφο Πίτερ Λίζε, τον εισηγητή και συμφωνώ με τις ε, παρεμβάσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει πραγματικά να επιδείξουμε σύνεση. Η ε, απόφαση της Επιτρόπου ήταν μια συνετή απόφαση, παρότι ξέρουμε ότι μια διεθνής συμφωνία για ένα τόσο δύσκολο ζήτημα είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Κύριος Πρόντι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Ήτρε καταψήφισα το backloading. Ακριβώς γιατί έχω την αίσθηση ότι αν επιλέξουμε ένα εργαλείο με γνώμονα την αγορά, θα πρέπει μετά να είμαστε ακόλουθοι στη στάση μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω και τη γνώμη μου, όλο και πιο αρνητική γνώμη, έναντι του πρωτοκόλου του Κιώτο. Ουσιαστικά, έχουμε φτάσει στο 15% των ε, εκπομπών Υπάρχουν χώρε λοιπόν που είναι στο 15% και είναι συνδεδεμένε ακόμα στο πρωτόκολλο του Κιώτο. Και πιστεύω ότι αν λάβουμε υπόψη τι δηλώσει στον Παλί που υπενθύμησε και ο συνάδελφο νωρίτερα, τότε πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση για το πρωτόκολλο του Κιώτο ένα ανανεωμένο πρωτόκολλο που θα πρέπει να περιέχει στοιχεία δικαιοσύνης και ισότητας. Σύμφωνα και με τη δήλωση του Μπαλί. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, της πολιτικής αεροπορίας, θέλω να το υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ιδίως σε ό,τι αφορά την χρήση του black carbon ε, από τα αεροπλάνα ε, στη στρατόσφαιρα. Γιατί στρατόσφαιρα αυτά τα μόρια του black carbon μπορούν, έχουν και θεκτικότητα να παραμένουν χρόνια. Στρατόσφαιρα, δηλαδή, όπου γίνονται και μετεωρολογικές αλλαγές. Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πραγματικά κατεπήγον ακριβώς λόγω του τρόπου τον οποίο αντιδρά ο άνθρακα στρατόσφαιρα. Ζητώ λοιπόν στη συζήτηση με τον ΙΚΑΟ να γίνει αναφορά και σε αυτή τη λεπτομέρεια. Διότι κατά τη γνώμη μου είναι λεπτομέρεια μεν, καθοριστική δε. Γιατί να πάρουμε μια απόφαση πέρα αυτού του περιορισμού. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. κάθε βήμα μπροστά που κάνουμε στη γνώση τελικά μας οδηγεί στην επιδίνωση ε, στο θέμα της υπερθερμής του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, να αξιοποιήσω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω τους εισηγητές και από την Επιτροπή Ένβη και από την Τραν για ε, τον ταχύτατο τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν για την εκπόνηση της έκθεσης αλλά και με το πόσο γρήγορα μελέτησαν τις ε, λεπτομέρειες της πρότασης. Ο αποφασιστικός τρόπος με τον οποίο εκπονήσαμε αυτό το καθήκον θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος ε, για μας γιατί εκφράζει την κατεύθυνσή μας και πώς ε, θέλουμε να εξελιχθεί ε, η διαδικασία ICAO. Τώρα, το κύριο στοιχείο της πρότασής μας είναι ότι είναι ε, πολύ λιτή η πρόταση γιατί είναι μια προσωρινή παρέκκληση του άρθρου 16. Δεν έχουμε αποδεχθεί ποτέ ότι θα αμφισβητηθεί η νομιμότητα της οδηγίας ETS, γιατί έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με την δική μας θέση σε ό,τι φορά την νομιμότητα της πρότασής μας αυτή, αυτός ο λιτός τρόπος ε, παρέκκλησης ε, από την οδηγία σε προσωρινή βάση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί και η ακαιρεότητα ε, της οδηγίας μας, του νόμου μας και για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνιμες στρεβλώσεις στον τομέα των αρωματοφορών και στους εμπορευομένους αυτού του κλάδου. Είτε αυτοί είναι Ευρωπαίοι είτε από τρίτες χώρες ε, αυτό το χρονικό όριο, το πολύ αυστηρό χρονικό πλαίσιο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Όμως, ε, σας καλώ αυτό το χρονικό πλαίσιο του ενός έτους να, ε, να προβληθεί και προς τα έξω, γιατί είναι κύριο στοιχείο της πρότασής μας. Ο ΙΚΑΟ ήταν και παραμένει ε, μια αφετηρία για μας ό,τι αφορά ε, τις ε, πολιτικές για την εμπορία εκπομπών. Με εκπλήσει όταν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κουμαντάρει όλο τον κόσμο, ενώ εμείς αναμφίβολα είμαστε βασικός φορέας εξέβρεσης λύσεων. Και είναι ένα ζήτημα, εμείς στηριζόμαστε στην εξωτερική μας ε, εικόνα και είμαστε περήφανοι για αυτήν. Και είναι δύσκολο και αποθαρρυντικό όταν βλέπουμε ότι κάποιοι εγκαταλείπουν αυτές τις ε, αρχές όταν είναι κάτι το οποίο έχει ε, προσδιορίσει την εικόνα μας προς τα έξω. Η συνολική αυτή προσέγγιση του ΙΚΑΟ αξίζει να, μια ευκαιρία. Είναι σαφέ ότι σε έναν ορισμένο, σε ένα συγκεκριμένο βαθμό όσοι αντιτίθενται στο ETS είναι ότι το ETS αποθαρρύνει την πρόοδο στο πλαίσιο ICAO. Τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, έχουμε ε, καταργήσει αυτή τη δικαιολογία των εταίρων μας να μην συμμετάσχουν στη συζήτηση που έχει ως στόχο να ε, καταλήξουμε σε μια λύση στην Ολομέλεια φέτος. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε με ειλικρίνεια ε, και ευθαρσός, αλλά και ως ε, άμεση ε, πρόσκληση προς τους εταίρους των τρίτων χωρών να μας δείξουν πραγματικά αν είναι διατεθειμένοι να καταλήξουν σε αποτελέσματα, να προσπαθήσουν. Και εμείς βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί τους. Για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και ξεκάθαρο τοπίο εδώ. Χρειαζόμαστε μια σαφή λύση που θα επιτρέπει στους εμπορευομένους ε, του κλάδου ε, να ενεργούν όπως προβλέπει η παρέκκληση. Όλοι οι εμπορευόμενοι ε, που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα έχουν τις ίδιες χρεώσεις και υποχρεώσεις. Επομένως, μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα υπάρχουν στρεβλώσεις και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού πρέπει να προστατεύονται βεβαίως. Κάτι τελευταίο για την διαδικασία του ΙΚΑΟ. Είναι σαφές ότι από το αποτέλεσμα αυτής της ε, διαδικασίας υπάρχουν ε, κατευθύνσεις εργασίας για την ομάδα ψηλού επίπεδου. Ε, οι προσπάθειες εξέβρεσης ενός κοινού πλαισίου που θα επιτρέψει την ύπαρξη διαφόρων NBM και αυτό είναι κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για την υιοθέτηση ενός ενιαίου NBM. Μετά έχουμε τις συζητήσεις ε, για το σφαιρικό και ολοκληρωμένο μέσο που προοδεύουν και θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Και τέλος υπάρχει και ένα τρίτο πεδίο ε, που αφορά μια δέσμη μέτρων, ε, διαφορετικών τεχνικών μέτρων. Και από πλευρά τη Επιτροπή είναι πραγματικά θεμελιώδου σημασία ε, τα αποτελέσματα που έχουμε στην διαδικασία της ΕΚΑΟ να προστατεύουν την περιβαλλοντική κυριότητα της πολιτικής μας. Και θα, το, θα το συνυπογράψουμε γνωρίζοντας με σιγουριά ότι έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα όπως το δικό μας ε, σύστημα ETS. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πέτερ Λίζο που είναι εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους για την ενθάρρυνσή τους. Γενικά ε, άκουσα υποστήριξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή Μεταφορών για την καλή συνεργασία και θα ήθελα να αναφερθώ ε, το θέμα του ανταγωνισμού ε, θα πρέπει να, ε, ο Ματιό Γκρός είπε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με, να λάβουμε υπόψη μας ε, ε, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αερογραμμών και νομίζω ότι το κάνουμε αυτό με την πρόταση αυτή. Δεν γίνεται διάκριση. Ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες ε, για ε, ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές ε, αερογραμμές. Εάν κάποια κινέζικη εταιρεία πραγματοποιεί πτήσει εντό τη Ευρώπης, τότε θα πρέπει να πληρώσει. Αντίστοιχα, αν μια ευρωπαϊκή εταιρεία κάνει μια πτήση εκτός Ευρώπης, δεν πληρώνει. Καθότι η τιμή για τα πιστοποιητικά ήταν αρκετά χαμηλή το 2012 ήδη, Ε, είναι Επειδή η τιμή ήταν τόσο χαμηλή, σημαίνει ότι δεν ισχύει το ε, επιχείρημα περί ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Θα πρέπει μακροπρόθεσμα να φροντίσουμε να βρούμε μια άλλη λύση ε, και γι' αυτό ε, η πρότασή μας περιορίζεται σε ένα χρόνο. Η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Ομπάμα, δεν απαγόρευσε από τις Αμερικανικές ε, εταιρείε να συμμετέχουν. Υπάρχει ένα διάταγμα ε, του Υπουργού, ε, αλλά υπάρχει περιθώριο διαπραγματεύσεων. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει ο Χόλκερ Κράμερ να διαβάσει την έκθεση. Ε, θα βρει απαντήσεις στα επιχειρηματά του. ο Μπάς δεν είναι παρόν. Α, είναι παρόν. ναι, θα μιλήσω αγγλικά. Καλά, θα μιλήσω γερμανικά. Ε, για πολιτικούς λόγους οι πράσινοι πρέπει να πούν ότι κρατάμε ψηλά τη σημαία και είμαστε οι μόνοι που ενδιαφερόμαστε για την προστασία ε, του ε, ε, περιβάλλοντος, αλλά σε παρακαλώ διάβασε το briefing των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα να κάνω έκκληση στην υπευθυνότητα των πρασίνων. Διαβάστε τι λένε οι εμπειρογνώμονες ε, του περιβάλλοντος. Συμφωνούν. Και ε, όσον αφορά αυτά που είπε η Κομισιόν, υπάρχουν δύο πιθανότητες ε, στην ΙΚΑΟ. Η πρώτη είναι η προτιμητέα λύση. Είτε θα βρούμε μια διεθνή λύση, τότε αξίζουν το κόπο οι προσπάθειές μας. Και εάν δεν βρούμε διεθνή λύση, τότε ο Μουτζούρης δεν ε, θα είναι πια στην Ευρώπη. Η Κομισιόν είπε να, ε, να, να καταργήσουμε τις δικαιολογίες. Ε, τους τελευταίους μήνες ε, και χρόνια ε, μιλώ με άλλες χώρες, τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα κλπ. Ε, που λένε ότι θέλουν διεθνή συμφωνία. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν θα υπήρχε διεθνή συμφωνία διότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Τώρα όμως είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν και αν τον Σεπτέμβριο δεν ε, έχουμε αποτελέσματα, τότε ε, δεν μπορούν πια να λένε ότι θέλουμε διεθνή συμφωνία, ε, διότι θα έχουν αποτύχει οι ίδιοι, οπότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε την οδηγία μας. Έχουμε λοιπόν μια διπλή ευκαιρία, ούτως ή άλλως θα ξεφορτωθούμε το Μουτζούρι και έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να πετύχουμε διεθνή συμφωνία, η οποία δεν θα είναι τέλεια, η οποία όμως θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του κλίματος και γι' αυτό αξίζουν τον κόπο οι προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πέτερ Λίζε, για, τα... για τις τελευταίες σου αυτές παρατηρήσεις. Η 28 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, ε, συζήτηση θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου, στις 26 Φεβρουαρίου. Θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και ενδεικτικά υπολογίζουμε με την Ολομέλεια του Απριλίου. Σφιχτό χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Ε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ε, θα τα ξαναπούμε στις 3 για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας.